ορίζεται λοιπόν και αυτή η εντολή. Τα πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση. Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις θα θεωρήσω και θα χορηγήσω, θα διαβιβάσω τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν σήμερα.